εδώ και δύο χρόνια ηγήθηκε της αποστολής στην Γεωργία. Ο πρέσβης Χάμπερ ήρθε εδώ να μας επισκεφτεί και πέρσι, λίγο πολύ την ίδια περίπου περίοδο, για να μας μιλήσει για αυτή την αποστολή, ειδικά. Έκτοτε ανέλαβε την ε, αρχηγία ο υπήν της CPCC, διότι είναι επικεφαλής των μη στρατιωτικών αποστολών που αποτελούν, αν θέλετε, και την μεγάλη πλειοψηφία των αποστολών που γίνονται στα πλαίσια της CPCC. Ε, η δομή αυτή είναι μια δομή η οποία τραβά την προσοχή της υποεπιτροπής μας, κύριε Πρέσβη, διότι τακτικά προβαίνουμε σε ακροάσεις και επισκέψεις στις διάφορες αποστολές. Και θα σας θυμίσω για ποια αποστολές, για ποιες αποστολές πρόκειται, αλλά όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει στις εκθέσεις μας, και πρόσφατα στην έκθεση του συναδέλφου Γκουαλτιέρη, ο οποίος φτάνει αυτή τη στιγμή, τα σώμεθα υπέρ και είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε η CPCC να έχει τα μέσα για να μπορεί να λειτουργήσει. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δομή και σε αυτή την περίοδο πλήρους αναδιοργάνωσης με τη δημιουργία αν θέλετε της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης η CPCC διαθέτει ειδικότερα τα μέσα σε προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει και ξέρουμε ότι τι εντάσει που ισχύουν και υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό είναι ένα ζήτημα πολύ λεπτό και ευαίσθητο για τι δομέ αν θέλετε σχεδιασμού και διεξαγωγή των επιχειρήσεων στρατιωτικών και μη. Ξέρουμε επίση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, ιδιαίτερα γρήγορο στην έκφραση δηλαδή και στην δημιουργία αν θέλετε ενό κοιτάρου, δηλαδή παγκοσμίου κοιτάρου, αν δηλαδή, σχεδιασμού και διεξαγωγή επιχειρήσεων στρατιωτικών ή πολιτικών επιχειρήσεων, μη στρατιωτικών δηλαδή, Πρόκειται για μια διαδίκηση παλαιά που είναι απολύτω λογική κατά την άποψή μα, ανάλογα με τι αποστολέ που χρειάζεται να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ωστόσο επίγνωση και των πολιτικών δυσκολιών που υπάρχουν σε επίπεδο Συμβουλίου, αλλά είμαστε πάντοτε προσιλωμένοι και θέλουμε η υπηρεσία εξωτερική δράση να διαθέτει μια τέτοιο κύτταρο γιατί ξέρουμε δηλαδή και τι πιθανέ αν θέλετε εικονικές αν θέλετε αποστολές που θα μπορούσαν να γίνουν Φερπίνη και να οργανωθούν σε περίπτωση τη Λιβύη, παραδείγματο χάρη. Όσον αφορά τώρα τι τρέχουσε αποστολέ τι οποίε θα ήθελα να σα υπενθυμίσω διότι είναι όλε τι πολύ σημαντικέ και πιο σημαντική είναι βεβαίω το Κωσυφοπαίδιο, αλλά έχουμε στο Αφγανιστάν, έχουμε επίση και στην Γεωργία, την οποία γνωρίζει και πολύ καλά, στην Βοσνία, UPM, ΕΠΟΛ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, εμπάμε Ραφά, στο Ιράκ επίσης, μια αποστολή που πολύ συχνά ξεχνούμε, στο Κονγκό επίσης, για την οποία θα έχουμε μια κρόση την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ των αποστολών αυτών, ορισμένες εξ αυτών, η εντολή προσεχώς εκπνέει. Θα πρέπει συνεπώ να γνωρίζουμε και θα θέλαμε να μάθουμε ποιε είναι οι απόψει όσον αφορά την συνέχιση ή αν θέλετε την αλλαγή, την τροποποίηση αυτών των αποστολών. Υπενθυμίζω πάντως ότι ο στόχος της ακρόασης δεν είναι να ξαναδούμε μία προς μία τις αποστολές αυτές. Θέλουμε να δούμε δηλαδή τις IPCC συνολικά, δηλαδή και την τοποθέτηση του αντέστου των θεσμικών οργάνων γενικότερα και το τι θα μπορούσε να την επηρεάσει με τη δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αν κάποιοι συνάδελφοι, και λογικό αυτό, έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα πάνω στι συγκεκριμένε αποστολέ, ο στόχο είναι να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια γενικότερη, αν θέλετε, πολιτική, αν θέλετε, εικόνα, σφαιρική εικόνα τη IPCC. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, η CPCC αποτελεί τμήμα των δομών διαχείρισης κρίσεων της ε, ευρωπαϊκής Εξωτερικής δράσεω στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας, το οποίο είμαι βέβαιος θα έχετε δει, βρισκόμαστε αν θέλετε στο πάνω δεξί μέρος. Και βρισκόμαστε στην, ε, στο Κόρτεμπεργκ Avenue, εδώ στις Βρυξέλλες. Όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν θα δούμε δηλαδή τις, ε, αποστολές που ορίζονται στις εξέλιξη, αλλά τις υφιστάμενες δομές Είμαι επικεφαλής αυτής της δομής για την οποία θα σας μιλήσω αλλά να αναφέρω επίσης και το πλαίσιο. Ποια είναι η θέση μας δηλαδή σε σχέση με τις άλλες δομές. Και πέρα στη CPCC έχουμε και την UMS για το στρατιωτικό προσωπικό και την διαχείριση, την διεύθυνση, την πολιτική διεύθυνση δηλαδή για διαχείριση των κρίσεων. και γύρω, γύρω τα θεσμικά όργανα για τα οποία εργαζόμαστε είναι η ΣΥΦΚΟΜ, την Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπή και βεβαίως και την πίεση. Και υπάρχουν και άλλα θεσμικά όργανα, ο ΣΕΤΣΕΝ και το ΡΕΧΟΝ επίσης, την European Defense Agency στη Μαδρίτη, μάλλον η European Defense Agency εδώ στις Βρυξέλλες διορθώνω και η UISS το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών τον, στο Παρίσι. Τι ακριβώς κάνουμε εμείς ως IPCC τώρα. Προερχόμαστε από την GD9 του Συμβουλίου, αλλά το 2007 όταν ήδη κάποιες πολιτικές αποστολές έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε ότι χρειαζόμασταν και ότι είχαμε ανάγκη μια πιο επαγγελματική αν θέλετε δομή προκειμένου να διεξάγουμε αυτές τις αποστολές. Και δημιουργήθηκε η PCC ως εκ τούτου. Έχουμε τώρα 8 αποστολές, 8. Έχουμε πραγματοποιήσει 15 τέτοιου αποστολές, επί συνόλου 23. Οι 8 υπόλοιπε είναι στρατιωτική, ήταν στρατιωτική φύσεω. Δεν υπάρχει αν θέλετε η μεικτή στρατιωτική και μη στρατιωτική δηλαδή επιχείρηση. Σημαντική εξέλιξη αυτή για το μέλλον. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει. Θα γνωρίζετε επίση και θα καταλαβαίνετε ότι η πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την άμυνα αναπτύχθηκε από τους ε, πολέμους, θα θέλετε, που ολοκληρώθηκαν ή τελείωσαν μάλλον με σημαντικό ρόλο βεβαίω του ΝΑΤΟ δηλαδή και των ΗΠΑ με στρατιωτικέ αποστολέ. Τα θεσμικά όργανα συνεπώ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο στρατιωτικό σκέλο ενώ οι περισσότερε από τι αποστολέ αυτέ στην οποία συμμετέχει δηλαδή, το ίμιση του προσωπικού γίνονται από την CPCC και είναι μη στρατιωτική φύσεω αυτέ οι αποστολέ. Τι κάνουμε τώρα επί καθημερινής βάσεως. λαμβάνουμε τι εκθέσει, πραγματοποιούν αυτέ τι αποστολέ, δηλαδή και λαμβάνουμε τι εκθέσει αυτέ, τι διαβιβάζουμε στη πίεση και στα άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία ενδιαφέρονται στην ημερήσια και την ημερήσια αν θέλετε διεξαγωγή των εργασιών αυτών και των παρακολουθούν την πορεία του. Αντιμετωπίζουμε επίση και κάποια επεισόδια, βλέπουμε τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να τροποποιηθεί. Μιλούμε με εκπροσώπους, αν θέλετε, της χώρας υποδοχής, ας πούμε έτσι, επισκεφτόμεθα τι αποστολέ για να αποκτήσουμε, θέλετε, έτσι και μια εκπρόσωπη όσους εντύπωση των όσων γίνονται εκεί. Επίση, στηρίζουμε τι αποστολέ αυτέ. Τι σημαίνει ανθρώπινη πόρη, χρηματοοικονομική στήριξη και κεφαλογικέ δαπάνε. Και το πιο σημαντικό όλων αυτών είναι βεβαίω η ανθρώπινη πόρη. Έχουμε προσωπικό 4.000 σε αυτές τις 8 αποστολέ συνολικά που συγκρίνεται με το προσωπικό δηλαδή άλλων μεγάλων θεσμικών ε, οργάνων που στέλνουν δηλαδή τέτοιου προσωπικό. 30.000 κοινωνικά και τα ένα έθνη. Βλέπετε ότι εμεί είμαστε σχετικά μικροί, για να μην μιλήσουμε τώρα για τον ΝΑΤΟ. και επίσης και του, της ΔΑΣΕ. Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο ενεργοποιούμεθα και είναι και τα θεσμικά όργανα με τα οποία, αν θέλετε, συναγωνιζόμεθα και ανταγωνιζόμεθα σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη, διότι όλα αυτά τα θεσμικά όργανα ε, είναι είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν, αν θέλετε, το απαραίτητο προσωπικό, δηλαδή στον ΟΑΣΕ, στον ΝΑΤΟ και πάει λέγοντα. Και χρειάζεται να έχουμε ε, επαρκές προσωπικό και βεβαίως η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών μια δεδομένη χρονική στιγμή είναι αποφασιστική σημασία αναφορικά και σχετικά με τον πόσο προσωπικό μπορούμε να, διαθέσουν, να μας διαθέσουν. Αυτό αποτελεί επίσης και συνιστά μεγάλη δυσκολία γιατί οι κρίσεις αυτές δεν εμφανίζονται αν θέλετε ταυτόχρονα με τον επιχειρηματικό κύκλο και με την εξέλιξη των οικονομικών δηλαδή των κρατών μελών ή τις εξελίξεις. Και ένα άλλο επίση πολύ σημαντικό αναφορικά με του ανθρώπινου πόρου, αν θέλετε, είναι τα προσόντα τα οποία έχουν. Θέλουμε δηλαδή εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί οι περισσότερου από αυτού που έχουν διάθεσή είναι αστυνομικοί. Και ξέρετε ότι μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ ενό του αστυνομικού, αν θέλετε, και προσωπικού των όπλων δυνάμεων είναι ότι οι στρατιωτικοί είναι πάντοτε διαθέσιμοι. Ενώ οι αστυνομικοί θα πρέπει αν θέλετε να εγκαταλείψουν τη θέση τους από την οποία θα λείψουν και βεβαίω τα κράτη-μέλη και τα Υπουργεία Εσωτερικών τα οποία εκφίσως δεν γνωρίζουν δηλαδή και τι γίνεται στον εξωκόσμο όπως τα Υπουργεία Εξωτερικών και τα Υπουργεία Άμυνας. Τα Υπουργεία Εσωτερικών δηλαδή διστάζουν να θέσουν τη διάθεσή μας αυτό το προσωπικό και απαιτούν συνεχείς επαφές μαζί τους προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους, πόρους, τους ανθρώπινους πόρους που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων είναι να έχουμε δηλαδή παρκές προσωπικό και κατάλληλα ειδικευμένο. Μέτρησα, μέτρησα βεβαίω. Αυτό το στοιχείο βέβαια δεν είναι και το σωστό γιατί τα, τα έτη του προπολογισμού δεν ε, αντιστοιχούν με τα έτη του προπολογισμού δηλαδή το ξένο action service ότι δαπανίσαμε γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή για τις δικές μας τις αποστολές δαπανώνται. Οι μερίσει αποζημιώσει που δίνουμε, δηλαδή σε εκείνου δηλαδή, του οποίου στέλνουν τα κράτη-μέλη, αποσπούν τα κράτη-μέλη, ο βασικό μισθό καταβάλλεται από το κράτο μέλο το ίδιο. Εμεί του δίνουμε αυτή τη μερίση αποζημίωση όπω κάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη και σε εκείνου δηλαδή του οποίου αν θέλετε είναι συμβαλόμενοι, δηλαδή προσωπικό, τα οποία τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να μα διαθέσουν, αλλά τα οποία εμεί θα πρέπει να προσλάβουμε, αν θέλετε, και να βρούμε δηλαδή στην ανοιχτή αγορά στην ελεύθερη αγορά μάλλον. Ένα άλλο σημαντικό σημείο της χρηματοδότησης είναι και ο εξοπλισμός. Και τα τεσσαρακισμένα οχήματα είναι το πιο σημαντικό. Και θα πρέπει να τα βρούμε αυτά τα τεσσαρακισμένα οχήματα εδώ στην Ευρώπη, την αγορά της Ευρώπης. Και βεβαίως αυτή είναι μια από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οι προμήθειες. Και οι προμήθειες αυτές διέπονται από τον χρηματοοικονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτός ο κανονισμός όπως ενδεχομένω θα γνωρίζετε, σχεδιάστηκε αρχικά για την κοινή αγροτική πολιτική, Φελιππίν ή για την αναπτυξιακή συνεργασία, την συνεργασία για την ανάπτυξη. Επομένως, έχει θέλετε και πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πιο μεθοδικό σχεδιασμό των δαπανών. Άρα μεγαλύτερες προθεσμίες από αυτές που συνήθως πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη μας για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και σε περίοδο κρίσεων. Και αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δυσκολία που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τη στήριξη αυτών των αποστολών. Κατόπιν και πέραν αν θέλετε τη καθημερινότητας όσον αφορά την διενέργεια αυτών των αποστολών Επίση κάνουμε και σχεδιασμό και μεθοδολογική ανάλυση. Βλέπουμε τι πρέπει να αλλάξει και τι μπορεί να αλλάξει όσον αφορά την εκπαίδευση αν θέλετε πρώτη ανάπτυξη δηλαδή του προσωπικού εκεί πριν δηλαδή να διενεργηθεί και γίνει αυτή η αποστολή. Τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε δηλαδή οικονομικά την αποστολή, πώς μπορούμε να θέλετε να την εκτιμήσουμε, να την ε, αξιολογήσουμε αυτή την αποστολή. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλέ φορέ, διότι η επιτυχία μιας αποστολή δεν εξαρτάται από την ίδια διαχείριση, αλλά και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εξωτερικά δεδομένα. Αν θέλετε, τα οποία αν θέλετε, μα δίνουν να θέλετε, οι εμπλεκόμενοι εκεί, επιτόπου δηλαδή που βρίσκονται σε σύγκρουση. Για τον λόγο λοιπόν αυτό η επιτυχία σε μεγάλο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζεται από εξωγενείς παράγοντες. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρηθεί πολλές φορές και να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα για το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η αποστολή ή τι δεν έκανε καλά ή τι δεν έκανε καλά η αποστολή αυτή ή δεν έγινε καλά στο πλαίσιο της αποστολής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θα κάνετε αυτή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποστολών. Και βεβαίως δίνουμε και συμβουλές αν θέλετε. Safecom για την Relex επίσης και στην PSC e, που είναι ο και βασικός μας πελάτης, ας το αποκαλέσω έτσι. Ναι. Τώρα ποιες είναι οι διαφορές στη διαχείριση των κρίσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα, το στρατιωτικό προσωπικό δηλαδή και σε MPD. Υπάρχει αν θέλετε πλήρης ασυμμετρία δηλαδή καθηκόντων σε σχέση με το στρατιωτικό προσωπικό. Διότι το στρατιωτικό προσωπικό σε αντιδιστολή με το δικό μας δηλαδή δεν διεξάγει αποστολές και δεν διενεργεί αυτές τις αποστολές. Ξέρετε δηλαδή τις συζητήσεις που γίνεται για τον πλήση και τα πλησιακά, το πλησιακό αν θέλετε στρατηγείο. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το στρατιωτικό προσωπικό αν θέλετε να έχει αν θέλετε, αυτό το αρχηγείο δηλαδή για να διεργεί τις αποστολές. Οι αποστολές αυτές γίνονται από τα εθνικά αρχηγεία δηλαδή, από το Potsdam δηλαδή. Αλλά οι Βρυξέλλες ακόμη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει, δεν της δίνεται γιατί της έχει δοθεί αυτή η άδεια και δεν της επιτρέπεται. Συμβουλεύουμε δηλαδή τη Στρατιωτική Επιτροπή και μόνο. Και η Στρατιωτική Επιτροπή με την συνέχεια συμβουλεύει δηλαδή τον είπα το πρόσωπο και την πίεση όσον αφορά τι στρατιωτικέ επιχειρήσει που πρέπει να γίνουν. Ο δικό του ρόλο δηλαδή είναι εντελώ διαφορετικό. Συμβουλεύουν και εμεί συμβουλεύουμε, αλλά διεξάγουμε επιχειρήσει κυρίω. Κατόπιν έχουμε και τη CMPD, την πολιτική διεύθυνση για τη διαχείριση των κρίσεων δηλαδή, με την οποία είχαμε και έχουμε πολλέ επικαλύψεις, διότι η CMPD ασχολείται επίση και με τι δικέ μα επιστολές, αλλά και με τι στρατιωτικέ. Η βασική διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι η CMPD ασχολείται με τις αποστολές κυρίως προτού να ξεκινήσουν. Επομένως, όταν εμφανίζεται κρίση και διαμορφώνεται συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει αυτή η αποστολή, τότε μπαίνει στο παιχνίδι η CMPD, τότε και μόνο, και αν θέλετε και φτιάχνει αυτό το σχέδιο αν θέλετε, διαχείρισης κρίσεως. Και βεβαίως συμμετέχουμε κι εμείς, διότι δεν είναι μόνο πολιτικής και στρατηγικής φύσεως η δουλειά αυτή. Ένα λεπτό, να απαντήσω στο τηλεφωνό μου. Εδώ Καμπούλ. Ε, Συμβουλεύουμε λοιπόν τη CMPD αναφορικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτοί φτιάχνουν, αν θέλετε, αυτή την, το concept δηλαδή για τη διαχείριση της κρίσης. Το Συμβούλιο αποφασίζει για την αποστολή αυτή και το επόμενο βήμα είναι εμείς επεξεργαζόμεθα ένα concept of operations και συμβουλεύουμε τον μελλοντικό επικεφαλή τη αποστολή αυτή για να φτιάξει τα σχέδια δηλαδή για αυτή την αποστολή. Όλα αυτά τα έχουμε δανειστεί από τον ΝΑΤΟ και τα έχουμε προσαρμόσει στι δικέ μα ανάγκε. Για τη μη στρατιωτική αντιμετώπιση κρίσεων δηλαδή. Όταν κάναμε την πρώτη αποστολή τέτοιου είδου στη Βοσνία το 2003 και θα κλείσει στο άμεσα προβλέψιμο μέλλον αυτή η αποστολή ή θα μειωθεί σημαντικά. Το 2003 δηλαδή δεν υπήρχαν άλλες διαδικασίες σχεδιασμού. Πέραν αυτών που είχε το ΝΑΤΟ. Επομένως τις πήραμε από το ΝΑΤΟ και τις προσαρμόσαμε στις δικές μας ανάγκες. Και μόλις διαχείριση της κρίσης και υπάρχουν και δομές στο Συμβούλιο αρχίζει η αποστολή. Όταν η αποστολή χρειάζεται να αλλάξει τη στρατηγική της κατεύθυνση τότε και πάλι μπαίνει στο παιχνίδι CMPD και συντάσσει μια στρατηγική αν αποτίμηση της αποστολής αυτής η οποία συζητάται κατόπιν GSE και αναλόγως αλλάζει η εντολή ή όχι. Ούτως όπως βλέπετε υπάρχει πολλή διάδραση με την CMPD Έχουμε και επικαλύψεις, αλλά είναι παραγωγικού χαρακτήρα αυτές οι επικαλύψεις. Αλλά δεν έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση με το στρατιωτικό προσωπικό, γιατί είναι μέχρι στιγμής καθαρά διαφορετικές οι αποστολές μας και έχουμε απλώς παροχή συμβουλών από αυτούς. Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλο δυναμικό, μεγάλες δυνατότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το να έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων στη διάθεσή της Μπορεί να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, μπορεί να κάνει πολιτικές επιχειρήσεις. Με όλα αυτά τα οποία κάνει η Κομισιόν λοιπόν και με την εργαλειοθήκη της ε, Κομισιόν μπορούμε να προχωρήσουμε και σε διαχείριση συγκρούσεων με πολιτικά μέσα. Εμείς έχουμε με το δικό μας σύστημα μια πολιτική αντιμετώπιση η οποία είναι σε συνεργασία με την Κομισιόν ώστε να υπάρχει μια συνοδευτική παρουσία μη στρατιωτικών μέσων και συγχρόνως έχουμε και μια στρατιωτική αποστολή. Πρέπει λοιπόν να ενοποιήσουμε την εργαλειοθήκη που έχει η Κομισιόν για τα θέματα αυτά και μία από τις προτάσεις είναι λεγόμενη πρόταση της Βαϊμάρης από τη Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία η οποία προτείνει ένα κοινό επιχειρησιακό στρατηγείο στην Λεωφόρο Κόρτεμπεργκ, όπου συναντιόμαστε και αλεπιδρούμε με τους στρατιωτικούς. Παραμένει βέβαια η αλυσίδα διοίκηση διαφορετική μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων της αποστολής και πρέπει να υπάρχει λόγω της φύσεως της ίδιας αποστολής αυτής διαφορετική διοίκηση, αλλά αλληλεπιδρούμε πολύ καλύτερα από ότι αν είχαμε απλώς μία αποστολή πολιτική που γίνεται από εμά και μία ε, εθνικά δικούμενη στρατιωτική επιχείρηση που εξαρτάται από τη δίκηση της Βρετανίας, της Γαλλίας ή της Γερμανίας κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν η οποία εκκρέμει αυτή τη στιγμή, το κατά πόσο θα εφαρμοστεί ή όχι. Ανεξάρτητα από αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους στενότερης συνεργασίας με το στρατιωτικό προσωπικό για να μπορούμε να προτείνουμε και να σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες αποστολές και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που από αυτή την άποψη είναι πολύ καλύτερο από αυτό που προσφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία για το πολιτικό τμήμα των αποστολών τους αυτό που γίνεται από τους ε, επιμέρους φορείς θα πρέπει να βασίζονται στην χρηματοδότηση ορισμένων χωρών. Προεξάρχουσα μεταξύ αυτών ομάδα χωρών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Θα ακούσω τα σχόλιά σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Πολλοί συνάδελφοι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Έχω και εγώ δύο ερωτήματα. Ένα είναι ένα θέμα σημαντικό και το οποίο το έχετε γνωρίσει και εσείς ως επικεφαλής αποστολής επί το οποίο η περίφημη αυτή δυσκολία που αναφέρατε σε σχέση με τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικού είναι φανερό ότι οι επικεφαλείς των ε, αποστολών, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους, της ενέργειάς τους, των χρημάτων τους για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο υλικό, τον εξοπλισμό. Προχωρούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση του να έχουμε κάπου ένα χώρο αποθήκευσης, ένα χώρο που μπορούμε να αποθηκεύουμε το υλικό μας. Μα τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί δουλεύει αυτό το μαραφέτη. Να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να έχουμε χώρο με ακούνη διερμηνής. λοιπόν, αυτή η υλική πλευρά, η πλευρά του υλικού που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των αποστολών, αν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα των ανθρωπίνων πόρων. Αναφερθήκατε προηγουμένως στι δυσκολίε που έχουν όλο και περισσότερα τα κράτη-μέλη για να θέτουν στη διάθεσή σας ιδιαίτερα προσωπικό το οποίο είναι ειδικευμένα στα δικαστικά και αστυνομικά θέματα γιατί πάντα υπάρχουν τα θέματα εσωτερικής πολιτικής που έχουν προτεραιότητα έχουν προτεραιότητα έναντι της διαθεσιμότητας αυτών των, ε, ε, αυτού του προσωπικού για αποστολές αυτού του είδους. Ποιο είναι το περιθώριο ελιγμών που έχετε εσείς ως επικεφαλής της ε, ΣΕΠΕΣΕΣΕ για τα ζητήματα αυτά. Εξαρτιόνται όλα από τους εκπροσώπους της ΚΟΠΣ ή παρόλα αυτά έχετε κάποιο περιθώριο ελιγμών για να μπορέσετε να έρθετε σε άμεση επαφή με ορισμένα υπουργεία. Και θα ήθελα να θέσω και το ερώτημα αυτό σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Έχετε πρόσβαση στα εθνικά κοινοβούλια, μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε τις εθνικές, ε, τα εθνικά κοινοβούλια πέραν της ΚΟΠΣ <clears throat> για την ανάγκη να υπάρχει ανθρώπινο υλικό και για τη χρησιμότητα των αποστολών που διενεργείται. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που θέλω να σας χθε. Ο Μιχαήλ Γκάλερ από το έλκα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην υποεπιτροπή μας. Και εγώ δεν ακούω πολύ καλά τον ήχο στην αίθουσα, αλλά λειτουργεί ακόμα η διερμηνία. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ντανζόν για τις προμήθειες. Επίση, θα θέλαμε να έχουμε αυτό το οποίο λέμε στα γερμανικά Zeughaus, ένα χώρο που τίθεται όλο το οπλοστάσιο, όλα τα υλικά. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ίσω αντί να έχουμε μεμονωμένε διαδικασίε προσφορών για κάθε ε, αποστολή, μήπω θα μπορούσαμε να έχουμε και μια συμφωνία πλαίσιο με ορισμένε επιχειρήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, να υπάρχει η πρόβλεψη για όλες αυτές τις ε, αποστολές και μέσα σε μια συμφωνία πλαίσιο να μπορεί κανείς να παίρνει υλικό από μια εταιρεία, να παίρνει αυτοκίνητα. Ε... Να είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Λοιπόν, να υπάρχει ένας κεντρικός χώρος αποθηκεύσης υλικού. Δεύτερον, αναφερθήκατε το πόσο δύσκολο είναι ιδίως στον τομέα της αστυνομίας, των αστυνομικών δυνάμεων, να βρείτε ειδικευμένους συνεργάτες από τα κράτη-μέλη για αυτές τις αποστολές. Και εδώ προστίθεται μια ακόμα προβληματική ότι και το ΝΑΤΟ καταβάλει προσπάθειες να δημιουργήσει πολιτικές δομές ή να μεταξελίξει κάποιες δομές γιατί θέλουν και αυτοί να έχουν μια πλήρη, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ε, νομίζω ότι όλο και περισσότερο το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα σας ενισχύσει αυτό ή όχι. Επίσης αναφερθήκατε στα θέματα των επιχειρησιακών ε, αρχηγείων για το τρίγωνο της Βαϊμάρης και η Πολωνική Προεδρία πιστεύω θα δώσει συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Ίσως ε, θα γίνει σαφές μετά και από την ε, κρίση της Λιβύης ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη για τέτοιο συντονισμό αλλά εσείς αναφερθήκατε ότι η οδό η οδός Κόρτεμπερκ γίνεται ένα είδο επιχειρησιακού αρχηγείου, αλλά εξακολουθείτε να εξαρτιέστε από τα εθνικά στρατηγία. Και γι' αυτό, κατά τη δική μου άποψη, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό <clears throat> η σχεδίαση να γίνεται με πιο πλήρη τρόπο από τις Βρυξέλλες. Ξέρω ότι οι Βρετανοί ε, απορρίπτουν μια τέτοια αντιμετώπιση, δεν θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός. Αλλά εξάλλου η κυρία Άστον θα μας φέρει τον Ιούλιο μια ενδιάμεση έκθεση. Εμείς θέλουμε όλοι να δούμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ενότητα και ολοκλήρωση στα θέματα αυτά. Αλλά βλέπω ότι αυτά τα οποία προτείνετε εσείς μάλλον έχουν τροχοπεδηθεί σε μεγάλο βαθμό. Eh Ευχαριστώ που ήρθατε καταρχήν. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου πιστεύουμε ότι θα έχουμε μόνιμη επαφή με τη στρατηγική αυτή δομή που είναι η CPCC. Όπως ε, υπενθύμησε και ο πρόεδρος Ντονζόν, αυτή η Επιτροπή και φέτος επεξεργάστηκε την ετήσια έκθεση για την ΚΠΑ, την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, με διάφορες προτάσεις. Μερικές από αυτές αφορούν το ρόλο, τη δομή της EPCC. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω σε αυτές τις προτάσεις και να τις συζητήσω μαζί σας. Καταρχήν, το Κοινοβούλιο διερωτήθηκε για την καταλληλότητα των πόρων, ανθρωπίνων πόρων της EPCC, σε σχέση με τα πολυάριθμα καθήκοντα και αρμοδιότητες που έχει. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα είναι ακριβώ αυτό. και τη διάσταση της του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έχετε ελάχιστος πόρους σε σχέση με τις πολυάριθμες αρμοδιότητές σας. Πέστε μου τη γνώμη σας για αυτό το σημείο, για το θέμα των ανθρωπίνων πόρων. Δεύτερον, για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών αυτών. Αυτό δεν υπάρχει στην έκθεση, απλώς από περίεργεια το ρωτάω. Από το οργανόγραμμα της EPCC βλέπω μια διαίρεση ανά αποστολή, όπου μοιάζει να μην υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό των ανθρώπων και στο μέγεθος αποστολής, μεγάλης, μικρής κτλ. Όταν εσείς αναλάβατε, ε, πιστεύετε ότι χρειάζεται ε, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το επίπεδο. Δεύτερον, η σχέση με την υπηρεσία της Κομισιόν, που διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό για τις αποστολές. Όπως θα είδατε στην έκθεση του Κοινοβουλίου, γίνεται μια πρόταση από το Κοινοβούλιο. Λάβαμε υπόψη μας και τη δουλειά που είχε γίνει από τον προκάτοχό σας στη PCC και αυτό που είχε πει η ίδια η Κομισιόν. Να εξορθολογιστεί δηλαδή αυτή η υπηρεσία αποστολών. Να δημιουργηθεί ίσως ένα γραφείο διαθεσμικό μεταξύ της CPCC και της Κομισιόν για να υπάρξει μια, ένας, μια συγκέντρωση κάποιων αρμοδιοτήτων και για να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο η απόκτηση σταθερών δυνατοτήτων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην χρειάζεται να απευθυνθεί στην αγορά κάθε φορά και τελικά να βρίσκεται με μέσα είτε λίγα είτε πολλά. Επομένω, να υπάρξει μια συγκέντρωση και διαδικασιών, να, έχουμε, να υπάρχει και προσωπικό συγκεκριμένο, να υπάρχουν και συγκεκριμένε σταθερέ δομέ. Τρίτο στοιχείο, το οποίο είπατε κι εσεί. Την συμμετρία μεταξύ της ασυμμετρία μεταξύ της ΕΠΣΣ και του στρατιωτικού προσωπικού. Αυτό το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι σημαντικό για, για μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει όμως τώρα μια νέα στάση από τους υπευθύνους της υπηρεσίας και από τα κείμενα του Συμβουλίου βλέπουμε ένα άνοιγμα ότι υπάρχει μια δυνατότητα, δηλαδή βαθμιαία τελικά, να βρούμε μια λύση. Ποια είναι η γνώμη σας για να απορροφηθεί αυτή η συμμετρία. Τέλος. Πειραματικά ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, λόγω της κρίσης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο αυτό που υπάρχει στην έκθεσή μας ε, Crisis Management Board, δηλαδή ένα συμβούλιο συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ε, επιχειρήσεων της ΚΠΑ Αυτή η προσπάθεια που γίνεται να συντονιστούν να συντονιστεί η διάσταση μεταξύ της ΠΑ και ο πιο γεωγραφικός ας πούμε, προσανατολισμός της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των υπολείπων φορέων. Ε, θα πρέπει να αποκτήσει πιο θεσμικό χαρακτήρα αυτό το board ή να γίνει πιο άτυπο. Έπειτα, το, το Κοινοβούλιο ε, συζητάει και θα ψηφίσει τον Ιούλιο τον δημοσιονομικό κανονισμό. Κάποιες από τις αλλαγές μπορούν να αγγίξουν και τη διαχείριση του προϋπολογισμού για τις αποστολές ε, μη στρατιωτικού χαρακτήρα, για τις πολιτικές αποστολές. Σκεφτήκατε αυτές τις προτάσεις, αξιολογήσατε αυτές τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και της εισηγήτριας Γκρέσλε. Μήπως θα υπάρξει μεγαλύτερη ακαμψία, ε, συμφωνείτε. Καλό θα ήταν να ακούσουμε από εσά τι πιστεύετε, γιατί θα μας βοηθούσε και εμάς. Είναι σημαντικό αυτό το έγγραφο, γιατί θα ρυθμίζει και τις, α, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο που ξοδεύονται αυτοί οι πόροι που διατίθενται. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Νικολάη. Έχετε ακούσει πολλές ερωτήσεις ήδη. Θέλω ήθελα παρόλα αυτά να σας κάνω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, ένα από τα βασικά καθήκοντα του μέσου σας. Και μια δεύτερη ερώτηση για τους ανθρώπινους πόρους. Τα κράτη-μέλη ετοιμάζουν, στέλνουν προσωπικό σε πολιτικές επιχειρήσεις. Εκπαιδεύουν τα κράτη-μέλη ή εκπαιδεύετε εσείς τα μέλη αυτά για τις αποστολές. Γιατί η ποιότητα των ανθρώπων αυτών είναι σημαντική για την επιτυχία των αποστολών. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Μια άλλη ερώτηση για τα κριτήρια πρόσληψης. Λαμβάνετε υπόψη σας τη διάσταση του φύλου τελευταία ερώτηση την ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε την αποστολή. Ε, θεωρείτε ότι στέφθη με επιτυχία η αποστολή στη Γεωργία. Bien. Euh, Πριν σας δώσω το λόγο κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας πω ότι έφτασε μια αποστολή από την Ινδονησία μόλις τώρα. National Resilience Institute που είναι ένα συντονισιακός φορέας όπου υπάρχουν και στρατιωτικοί και μη στρατιωτικοί ψηλού επίπεδου οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεξάγουν μια αποστολή ε, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα στις Βρυξέλλες. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Στην υποεπιτροπή μας λοιπόν έχουμε και τον πρέσβη, τον κύριο Χάμπερ που είναι δίπλα μου, ο οποίος είναι επικεφαλής της EPCC στη δική μας ιδιόγλωσσα. Να σας το πω στα αγγλικά που είναι το Civilian Planning and Contact Capability της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το άτομο που είναι επικεφαλής ε, όλων των αποστολών ε, μη στρατιωτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε οκτώ αποστολές ε, σε όλο τον κόσμο που διεξάγει αυτό ο φορέας. Αυτά τα λέω και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις προς τον πρέσβη και μετά να ακούσουμε και μια παρέμβαση από την Ινδονησιακή Αντιπροσωπεία, ο πρέσβης. Ευχαριστώ. Θα διεξέλθω με τη σειρά τα ερωτήματά σας η αποθήκη υλικού, <clears throat> ο χώρος αποθηκεύσης του υλικού. Αυτό θα επετάχυνε την ταχεία ανάπτυξη, φυσικά. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αποστολές μας αναπτύχθηκαν κάπως βραδέως στο κοσμοπέδιο χρειαστήκαμε ένα χρόνο προετοιμασίας, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ ταχύς αναπτύξεις όπως έγινε στην Γεωργία. όπου χρειαστήκαμε μονάχα δύο εβδομάδε μετά την απόφαση του Συμβουλίου. Τα πράγματα πήγαν από, από τα εξωτερική άποψη καλά, αλλά στο εσωτερικό υπήρξαν πολλές τριβέ, πολλά σημαντικά στοιχεία δεν είχαν ακόμα ε, συλλεγεί, δεν είχαν αγοραστεί όταν εγώ έφυγα από εκεί, ιδίως στον τομέα εσωτερικής ασφαλείας. Το να υπάρχει λοιπόν ένας χώρος αποθήκευσης αυτό θα βοηθούσε, βέβαια θα οδηγούσε και σε κεφαλαιουχικό κόστος. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αυτή η ιδέα της αποθηκεύσης, η εναλλακτική λύση που αναφέρεται κύριε Γκάλερ, να υπάρχει μια συμφωνία πλαίσεων για βασικά στοιχεία που πρέπει να ε, αποτελούν το υλικό, να υπάρχουν παραδείγματος χάρη υπολογιστές, ε, υλικό επικοινωνίας, τεθωρακισμένα οχήματα. Αυτό το κάνει η Κομισιόν ήδη από την εποχή που έγινε η ανάπτυξη της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γεωργία. Υπήρξε μια συμφωνία πλαίσιο όταν έγινε αυτή η ανάπτυξη για τεθωρακισμένα οχήματα. Αλλά η εταιρεία η οποία ήταν ο ανάδοχος Επτόχευσε και δεν μπορούσε να μας δώσει τα οχήματα αυτά. Και αυτό σχεδιάσαμε με πολλά οχήματα διαφορετικών χρωμάτων και προελεύσεων. Αυτό δυσκόλεψε την αποστολή και υπήρξε και ένα θέμα για την ασφάλεια της αποστολής. Κανονικά τα οχήματα αυτά είτε είναι του, της, του ΟΑΣΕ ή των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον θα πρέπει να είναι λευκά για να είναι αναγνωρίσιμα. Έκτοτε λοιπόν υπήρξαν πολλές άλλες συμφωνίες πλαισίου, αλλά δυστυχώς μόνο μετά από την απόκτηση αυτών των στοιχείων υλικού βάσει της κειμένης διαδικασίας. Καμία λοιπόν από αυτές τις διαδικασίες δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες, ούτε και αυτή για τα, εκτός από αυτή για τα τεθωρακισμένα οχήματα. Το κόστος λοιπόν το πολιτικό του να ξεκινάει κανείς μια επιχείρηση ταχεία ανάπτυξη και να μην μπορεί να κάνει μια ταχεία ανάπτυξη, το κόστο για μια τέτοια αποστολή, αν αστοχήσει, είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό προτιμούμε την επιλογή του να έχουμε μια αποθήκη υλικού. <clears throat> για το προσωπικό τώρα. Ιδίω για τα δικαστικά και αστυνομικά θέματα. Κάνουμε προσκλήσεις για συνεισφορές προς τα μελη μέσα από την κόψη. Θα περάσει μετά αυτή η αίτηση στις ε, εθνικές αρχές, στα εθνικά υπουργεία, που θα πρέπει βέβαια να περάσουμε σαν από τις επιχειρησιακές δομές μέχρι τα επίπεδα αυτών οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Τα ενδιάμεσα στελέχη βέβαια δεν χαίρονται ιδιαίτερα για τέτοιες <clears throat> αιτήσεις συμβολής και υπάρχουν τριβέ για αυτά τα θέματα. Γνωρίζω ποιε είναι οι συνθήκε στη χώρα μου, στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα θέματα αυτά. Έχουμε ομοσπονδιακή αστυνομία, έχουμε αστυνομία στα Λέντερ, έχουμε μια κλίδα κατανομή, ε, κάποια κρατήδια δεν συμμορφώνονται, έχουν ε, δυσκολίε χρηματοδότηση. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ βέβαια έχω αναλάβει τα καθήκοντά μόνο πριν από δύο μήνες θα προσπαθήσω <clears throat> να εξασφαλίσω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών μας από τις εθνικές αρχές, αλλά θα παραμείνει ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν υπάρχει έλλειψη θέλησης από την πλευρά αυτών οι οποίοι θα αποτελέσουν τα μέλη των αποστολών στο μέλλον. Προτιμάτε να έχετε πεπειραμένους στις ε, αποστολές αυτές, αλλά η ενδιάμεση <clears throat> ε, επικεφαλής τα θέματα χρηματοδότησης ε, και τα νομικά προβλήματα, όλα αυτά είναι μια τροχοπέδη στα θέματα αυτά και έχουμε και τους ανταγωνιστές μας. Ο ΑΣΕ, Ηνωμένα Έθνη, ΝΑΤΟ. Και αναρωτιέμαι, αλλά αυτό να πρόκειται σε εσά να αποφασίσετε, μήπως την περίπτωση αυτή να μην έχουμε μια προσέγγιση πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τις αποστολές μας πιο αποτελεσματικές. ώστε η πολιτική συνιστός του ΝΑΤΟ το ΝΑΤΟ βέβαια έχει κάθε δικαίωμα να υιοθετήσει μια δική του ολοκληρωμένη στρατηγική. Αλλά είναι προφανές, ήταν προφανές εδώ και πολύ καιρό, ότι οι στρατιωτικές αποστολές πρέπει να έχουν και μια πολιτική συνιστός. Αυτό είναι μια μεθοδολογία που έχει αναγνωριστεί σε όλες αυτές τις αποστολές. Το ερώτημα και πάλι είναι, <clears throat> εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των μελών του ΝΑΤΟ, σε ποιο βαθμό θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πορεία. Και όπως είπα προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αντί του ΝΑΤΟ, έχει πολλά βέβαια μειονεκτήματα, κλίμακα σχεδίασης, η πόροι του ΝΑΤΟ είναι αχανή σε σχέση με αυτού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά με την εργαλειοθήκη της Κομισιόν, με όλα τα πολιτικά εργαλεία σχεδιασμού, εμείς μπορούμε να έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων για να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσει από τη στρατιωτική μέχρι την πολιτική πτυχή. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν αυτή την ε, επιλογή και να προωθήσουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και να αφήσουμε τα κατημέλια να δίνουν περισσότερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στο ΝΑΤΟ. Κόρτεμπεργκ τώρα έναντι εθνικών ε, αρχηγείων. Γιατί υπάρχει αυτή η συμμετρία. Είναι παλιά η συζήτηση. Ε, ήδη την κάναμε στην δεκαετία των 90. Um, uh, το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά δεν θέλει να κάνουμε τα ίδια με το ΝΑΤΟ. Και υπάρχει και το θέμα του, της αποτελεσματικότητας και του κόστους. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το επιχείρημα. Αλλά τελικά εξάρτηται από τα κράτη-μέλη, όχι από μένα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα ήταν σημαντικό πλεονέκτημα αν είχαμε ένα αρχηγείο γιατί ο συντονισμός ε, είναι δύσκολος και όσο πιο μακριά είμαστε οι μένα τους δε, τόσο πιο δύσκολο να συντονιστούμε. Νομίζω ότι αν έχουμε και τις δύο διαστάσεις, ε, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές, ε, αυτό το αρχηγείο θα βοηθήσει και το συντονισμό καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Πόσο επαρκής, ε, ρώτησε ο κ. Γκουελτιέρη, είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Είναι καλά τα στελέχη. Και όταν πάνε επί τόπου, αναπτύσσουν ικανότητα να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Αλλά φυσικά, από όλους τους ανθρώπινους πόρους μας υπάρχουν διαφορές, ασυμμετρίες. Είναι διαφορετικά προετοιμασμένοι, διαφορετικά τους προετοιμάζουν τα κράτη-μέλη. Για την ποσότητα ρώτησα, λέει ο Υπάρχει ένα δίλημα προφανώς. Απ' τη μία υπάρχουν, υπάρχουν τα Υπουργεία Οικονομικών και απ' την άλλη έχουμε τις κρίσεις. Υπάρχει αυτή η διελκυστίντα. Δεν κινούν. Εμείς ανταγωνιζόμαστε για περισσότερους ανθρώπινους πόρους, αλλά λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο ανεπαρκών ε, οικονομικών πόρων. Μα πιέζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το επιλύσουμε όσο θα βασιζόμαστε εδώ. Αν μπορούσαμε να προσλάβουμε από την αγορά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά τότε το κόστος αυξάνεται. Και θα έπρεπε να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να προσλάβουμε πέρα από αυτό που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Φυσικά το πλαίσιο το θέτει ε, η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών και αυτό το αισθανόμαστε έντονα καθημερινά. Τώρα, η σχέση ανάμεσα στο προσωπικό της EPCC και τις αποστολές. Έχουμε 60 μέλη, η CMPD έχει 70 και 180 ε, οι στρατιωτικέ αποστολέ. Μπορεί να ξέρετε αυτά τα νούμερα. Δεν αρκούν 60 άτομα για να αντιμετωπίσουμε τις 8 αποστολέ μας. Φυσικά, οι στρατιωτικοί κάνουν του υπολογισμού τους υπολογισμούς τους και λένε ότι ένα αρχηγείο μπορεί να διαχειριστεί 120 αποστολές. Αλλά φυσικά κάθε στρατιωτικό θα σα δώσει άλλο, άλλη απάντηση. Στις δικές μας αποστολές, το αρχηγείο είναι τμήμα της αποστολής. 120 αν είναι συνήθιση η αποστολή, αλλά έχουμε 8 τελείως διαφορετικές αποστολές. Έχουμε διαφορετικά προβλήματα, διαφορετική εμβέλεια σε κάθε αποστολή, δεν ακούν αυτά τα άτομα ίσα ίσα που τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε χάρη στην αφοσίωση των μελών. Ε, στο Κοσμοπέδιο έχουμε τη μεγαλύτερη αποστολή. Και έχουμε τρία άτομα εκεί. Τρεις υπαλλήλου. Είναι πάρα πολύ καλή, Ευτυχώς και τα καταφέρνουν. Αλλά μόλις φύγει ο ένας, μόλις μετατεθεί, ο χαρτόπυργος αυτός θα καταρρεύσει το λέω αυτό στους δικούς μου μάνατζερ, δεν αρκεί το προσωπικό. Έχουμε και το υποστηρικτικό προσωπικό των Βρυξελών για τις αποστολές. Είναι μέλη που δουλεύουν στις Βρυξέλλες, μέλη αποστολών, για να διευκολύνουν θέματα προμήθειας. Αλλά εμείς πρέπει να τους τακτοποιήσουμε, πρέπει να τους κρατήσουμε ως μέλη της EPCC για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις αποστολές. Αυτό σημαίνει ότι τα, τα τακτικά μας μέλη, δηλαδή οι υπάλληλοι μας, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν, να αυξηθούν. για τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, το ξέρετε. Αλλά τώρα α, η αρμόδια υπηρεσία είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Συνομιλούμε μαζί του και για το θέμα τη αποθήκη υλικού και για αυτό το κοινό κέντρο υπηρεσιών, αν σα κατάλαβα. Ω πρώην επικεφαλή αποστολή έχω μια εμπειρία που με βοηθάει και πιστεύω ότι αυτέ οι δομέ θα πρέπει να είναι τμήμα τη EPCC και να μην είναι διαθεσμικές. Δεν θέλω να μειώσω τον έλεγχο και την εποπτεία τη Κομισιόν που είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό και τον δικό μα προπολογισμό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και έλεγχο από την Κομισιόν, αλλά ξέρουμε τι ανάγκε των αποστολών καλύτερα, γιατί ταξιδεύουμε συνέχεια, συνομιλούμε τηλεφωνικά με τα άτομα που είναι εκεί, ξέρουμε τι χρειάζονται. Και τη στιγμή που υπάρχει η CPCC ανάμεσα στην αποστολή και στην σε, μια, σε ένα διαγωνισμό πούμε, για προμήθεια, μπορεί, μπορεί ας πούμε, εμείς ξέρουμε τι, τι, χρειάζεται και αν πάει κάτι στραβά εμείς το ξέρουμε. Και θα πρέπει με αυτό το κέντρο να εξασφαλίσουμε και την εγκύτητα, α, τη δική μας απέναντι στις αποστολές, αλλά και να εξασφαλίσουμε και τον έλεγχο και την εποπτεία από πλευράς κομισιών. Πιστεύω ότι εκεί είναι το έλλειμμά μας. Εκείνο το έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Αποστολής σε σχέση με τις αποστολές του ΟΗΕ και της ΟΑΣΕ. Όταν ήμουν στη Γεωργία υπήρχε μια αποστολή του ΟΗΕ και, του, και της ΟΑΣΕ και μπορούσαμε να συγκρίνουμε. Πήραμε πολλά, πολλούς υπαλλήλους από αυτούς. Ε, και δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Πήγε πολύ καλή η αποστολή UMM, μόνο το θέμα της προμήθειας δεν πήγε καλά. Επομένως, ένα πιο κέντρο είναι βασικό στοιχείο για να δουλέψει η... καλά η αποστολή και το άλλο είναι το... η ανθρώπινη πόρη. Για τις προτάσεις στην έκθεσή σας. Αυτούς τους δύο μήνες που είμαι στη θέση αυτή, ομολογώ, αναγνωρίζω ότι δεν είχα το χρόνο να τα διαβάσω και να τα χωνέψω. Πρέπει να καθυστερήσω τις απαντήσεις και να σας τις δώσω στην επόμενη παρουσία μου, στην επόμενη επίσκεψη στην Επιτροπή σας. Απάντησα? Μπορείτε να απαντήσετε αυτό που θέλετε να απαντήσετε, αυτό που μπορείτε να απαντήσετε. Είστε ελεύθερος. Για την κυρία Νικολάη, η κατάρτιση για τα μέλη της αποστολής. Φυσικά κάνουμε μια αρχική εκπαίδευση για να εξοικειώσουμε τον κόσμο με τον τόπο κτλ. Μερικές φορές το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να σέβεσαι το πλαίσιο ασφάλειας τη αποστολή από την πρώτη μέρα που φτάνεις εκεί. Ε, υπάρχουν πολλές τοπικές συνθήκες, ε, πολιτιστικές διαφορές και οι σχέσεις των φίλων, πούμε, σε χώρες όπως το Αφγανιστάν ή το Ιράκ είναι πολύ σημαντικές. Φυσικά κάνουμε μια κατάρτιση πριν πάει το άτομο επιτόπου. Κάποια κράτη έχουν τέτοια κατάρτιση, η Σουηδία, Φιλανδία και Γερμανία κυρίω, αλλά άλλε χώρε μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατάρτιση. Υπάρχει παρόλα αυτά ε, συνολικά μια τεράστια ασυμμετρία σε αυτή την κατάρτιση πριν ξεκινήσει κανεί την αποστολή. Με αυτό ασχολούμαστε και στην CPCC. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα γιατί προσλαμβάνουμε κόσμο και ε, μόλις έρθει σε εμά, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει τον άτομο αυτό να το στείλουμε στην αποστολή πάρα αυτά. Και οι χώρε τους, από τις οποίες θέλουν, αποσπάτε, ξέρω εγώ, ή τον στέλνουν, τον αφήνουν τελευταία στιγμή. Εμείς θέλουμε να τον εκπαιδεύσουμε. Από την άλλη, θέλουμε να είναι και αποτελεσματική αποστολή. Δεν έχουμε πολλά ε, οικονομικά, οικονομικούς πόρους. Όταν, παραδείγματο χάρη, φτάνει κάποιο και έχει μία εβδομάδα για να εκπαιδευτεί, ο προκάτοχό του έχει ήδη φύγει. Κρίμα είναι, ίσω θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε αυτό το στοιχείο. Η κατάρτιση πάντως είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Τα κριτήρια για την πρόσληψη. Για το αποσπασμένο προσωπικό. Παραδείγματο χάρη πρώην αστυνομική. Ε, επιλέγουν εδώ τα κράτη-μέλη ουσιαστικά. Αλλά για τους, για τους managers έχουμε διαδικασία επιλογής για τα διευθυντικά στελέχη. Θα την ξέρετε γιατί περίπου είναι ίδια με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Με συνεντεύξεις κτλ. Η Γεωργία ήταν επιτυχής αποστολή. Εδώ θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά έτσι σύντομα μπορώ να σας πω η αποστολή έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Νομίζω τώρα πρέπει να αναπτύξουμε μια πολιτική για τη γεωργία. Και η μετάβαση αυτή είναι δύσκολη πάντα. Από μια αποστολή δηλαδή στην ανάπτυξη πολιτική, στη δημιουργία πολιτική. Γιατί ε, συχνά η αποστολή μοιάζει με υποκατάστατο τη πολιτική, αλλά δεν είναι υποκατάστατο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρέσβη. Δύο τελευταία ερωτήματα. Ο κύριος Βάγκελ. Αν αυτή τη θέση τη λάβει κάποιον που έχει αν θέλετε εμπειρία και από τη σημερινή συζήτηση κύριε Πρέσβη κατάλαβα ότι μιλάτε εκ πείρας. Μιας όμως και βρεθήκατε και εσείς στη Γεωργία θα ήθελα να διευρύνω κάπως τη συζήτηση και να σας θέσω και μια ερώτηση. Υπάρχει πραγματικά ανάγκη, υπάρχει προστιθέμενη αξία, εάν είχαμε αποστολή στον Αργόνο Καραμπάχ, δεν έχουμε μια τέτοια αποστολή του είδους αυτού στον Αγκόρο Καραμπάχ ακόμη δεν ξέρω βεβαίως και ποιος ε, αν υπάρχει ρόλος αν θέλετε και για αποστολή του ΟΑΣΕ αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό υπάρχει αυτό το αδιέξοδο παρά βεβαίως τις αισιόδοξε εκθέσεις που ακούμε από καιρού εις καιρών αλλά αυτό ήταν το ερώτημά μου τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον δεν εκπροσωπούμεθα στην ομάδα του Μίνσκ, πράγμα το οποίο είναι λάθος. Και κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία το κριτικάρω αυτό. Διότι νομίζω ότι θα πρέπει να μας εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αποστολή στον Αγκόρο Καραμπάχ. Και το δεύτερο ερώτημά μου αφορά το checkpoint θέση Ράφα. Από ό,τι γνωρίζω από τις 11 Μαΐου δεν έχουμε κανέναν εκεί. Ή παρετάθη. Στην Λορέα της Γάζας, έτσι. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον πρέσβη Χάμπερ για την παρουσίασή του. Νομίζω για πρώτη φορά κατάλαβα τι βρίσκεται πίσω από το ακρονίμιο CPCC. Και γνωρίζω επίσης ότι δεν υποτίθεται ότι μπορούμε να συζητούμε όλες και να συζητήσουμε σήμερα όλες τις αποστολές μία προς μία. Αλλά να ενισχύσω αυτό το οποίο είπε η πρώτη Νικολάη σχετικά με τη Γεωργία. Λίγη εντολή Σεπτέμβριο φέτος και σε ό,τι αφορά τη νέα εντολή ή μια νέα εντολή, πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Εγώ θα μπορούσατε να μα πείτε αν θέλετε αυτή η νέα, αν θέλετε αποστολή, αν θέλετε τι εντολή θα έχει. Και ο Άντρε τη σκέψη θα συνεχίσει ή θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον που θα έχει εκπαιδευτεί εκ των προτέρων. Άκουσα επίση για την ιδέα συγχώνευση των εντολών του εκπροσώπου για τον Νότιο Κάφκο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δηλαδή και με εκείνο δηλαδή για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Γεωργία και αν ναι τότε ο επικεφαλής της, παρακολούθηση ε, παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής θα συνδεθεί με τον νέο αν θέλετε εκπρόσωπο, τον δικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τον Αγκόνο Καραμπάχ. Αυτό αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ και πάντα σε όλες αυτές τις ε, συγκρούσεις υπάρχουν φυσικά θεσμικοί ανταγωνισμοί μεταξύ φορέων όπως ο ΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι δυνητικοί πάροχοι αποστολών. Τώρα για την γεωργία που αναφέρατε, μην μου περιμένετε να σας πω κάτι για το Ναγκόνο Καραμπάχ. Από την εμπειρία μου στη Γεωργία είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Η Αυχασία και το Ναγκόνο Καραμπάχ, παραγωγικά και η Οσετία έχουν πολύ μικρές, πολύ λίγη σχέση μεταξύ τους. Πολύ μικρή συγκρισιμότητα. Αν είχαμε βέβαια μία εντολή θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία αποστολή στον ναγκονο Καραμπάχ αλλά και ο ΑΣΕ θα ήθελε να το κάνει αυτό τώρα. Κατά πόσο θα τροποποιηθεί η δομή της ομάδας του Μίνσκ και η εντολή της θα ήταν κάτι το οποίο σε άλλους εναπόκειται, αλλά μια αποστολή στον Αγκόνο Καραμπάχ θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από αυτή στην ε, Γεωργία. Όπως ξέρετε υπάρχουν ένοπλες σειράξεις ε, σε καθημερινό επίπεδο. Το Αζερμπαϊτζάν επανεξοπλίζεται. Η ανησυμετρία μεταξύ των δύο χωρών Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν γίνεται πιο έντονη. Φοβούνται πολύ οι πυρογνώμες ότι μπορούσε να ξεσπάσει ένα πόλεμο μεταξύ των δύο κρατών. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε λοιπόν μια αποστολή, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από πολιτικέ κρίσει που πρέπει να γίνουν σε άλλα επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το ράφα, το πέρασμα της ράφα, συγγνώμη, Έχουμε φύγει από το 2007, όταν μας αντικατέστησε η Χαμάς. Εφόσον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και εφόσον το να μείνουμε στην περιοχή της, του σταθμού διέλευσης της Ράφα θα σήμαινε de facto συνεργασία με τη Χάμας, είμαστε υποχρεωμένοι να μην έχουμε ενεργή αποστολή. Η αποστολή αυτή έχει μειωθεί λοιπόν σημαντικά σε αριθμό ατόμων είναι αδρανής αλλά είναι και ο, ε, έχει χαρακτήρα ε, τρίτη, τρίτης ε, πλευράς που έχει το δικαίωμα να παρίσταται μετά από τη συμφωνία του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους. Αν φύγει η αποστολή από εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένα κενό. Και γι' αυτό κρατάμε την αποστολή επιτόπου σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, κάτι το οποίο έχει δώσει να βγει σε επικρίσεις. Αλλά εγώ έχω πάει πρόσφατα εκεί και η Ισραηλινή πλευρά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία προοπτική για την ε, αναζωγόνηση αυτής της αποστολής μας είπανε ας μείνετε τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου. Ένα πρόκειται λοιπόν στην ε, πολιτική ε, σχεδίαση να αποφασίσουν για το θέμα αυτό τους υπεύθυνους της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η εντολή για τη Γεωργία μάλλον θα παραταθεί για κάνα χρόνο ακόμα μετά από τις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε εκπνει εκπνέει κανονικά, γιατί υπάρχει τακτική παράταση κατά ένα χρόνο αυτής της εντολής και ο στρατηγός του Σκέβιτς, ο νέος αρχηγός αποστολής δεν είναι ακόμα εκεί, θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 18 Ιουλίου, νομίζω. Και μετά η εντολή του θα τρέξει τουλάχιστον μέχρι την αρχή της επόμενης περίοδου. Μετά το Σεπτέμβριο δεν θα μείνει μόνο για δύο μήνες, αυτό είναι φανερό. Νομίζω ότι αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάτι. Τι παρέλειψα. Ah, uh, Οι δύο USR έχουν συγχωνευτεί επίσης. Η νέα συγχωνευμένη ε, οντότητα θα είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα του Καυκάσου. Όταν εγώ ήμουν υπεύθυνο εκεί είχα επαφή και με τι δύο συνιστώσει USR που υπήρχαν όπω και με την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ω αρχηγός αποστολή συμμετείχα και στι διαπραγματεύσει τη Γενέβη που ήταν στις οποίες συμμετείχε μία από τις δύο USR. Μια πολιτική απόφαση είναι αυτή. Η ύπαρξη αυτών των EUSR κάνει πιο δύσκολο για τις αντιπροσωπείες να αναπτύξουν πολιτική εμπειρογνωμοσύνη. Γιατί όσο υπάρχει μια EU, EUSR θα είναι πάντα ο προτιμόμενος συνομιλητής της ε, κυβερνήσεως της χώρας στην οποία βρισκόμαστε ενώ ο αρχηγός της αντιπροσωπείας είναι μονάχα υπάλληλο τους, υποκείμενος τους. Αυτό δυσκολεύει λοιπόν την προσπάθεια να έχουν αρκετή ικανότητα όλες οι αποστολές σε επίπεδο πολιτικών συμβούλων. Οποιαδήποτε όμως αποστολή στην Γεωργία θα πρέπει να είναι σε μεγάλη και στενή επαφή με τις EUSRs. Είναι ένα δύσκολο και σημαντικό έργο να μπορεί να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας ενιαίος παίκτης η αντιπροσωπή από μια μεριά και η αποστολή από την άλλη πλευρά. Γιατί η αντιπροσωπεία δίνει απτά ωφέλη σε μια χώρα όπως είναι η διευκόλυνση για τις προξενικέ θεωρήσεις, η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά να υπάρξει και κάποια πολιτική ανταπόδηση. Αν λοιπόν <clears throat> ε, ενοποιήσετε αυτές τις δύο δομές θα υπάρχει σύγκρουση σε ορισμένα σημεία. Αν τις καθίσετε χωριστά, μπορείτε να δίνετε κάτι με το ένα χέρι και να το παίρνετε με το άλλο. Αλλά δεν μπορείτε να το παίρνετε με το άλλο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συντονιστούν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ρωτήσατε στην αρχή για το CPCC. Εντάξει. Τότε έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Νομίζουμε ότι έχετε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Νομίζω ότι μας κάνατε μια πολύ καλή επισκόπηση, όπως είπε και ο κύριος, κύριος Ταράν. Η δομή επί της οποίας υγείστε δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να την παρουσιάσετε ενδελεχώς στη λειτουργία της και στη δομή της. Νομίζω ότι έχετε <clears throat> ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Θα θέλαμε να σας υποδεχόμεθα πιο τακτικά με τους επιμέρους επικεφαλής των Αποστολών και πιστεύω ότι από τις 12 Ιουλίου θα σας ξαναδούμε όταν μιλήσουμε και για την πολιτική και την στρατιωτική μας ε, αποστολή στο Κονγκό η οποία έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα στους βουλευτές. Στις 12 Ιουλίου λοιπόν θα, έρθουμε, θα σας συναντήσουμε και πάλι να μιλήσουμε το Κονγκό. Κατά τα άλλα σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε καλή ανάληψη καθηκόντων γιατί όπως είπατε ακόμα είσαστε στη διαδικασία ανάληψη καθηκόντων σας. Και καλό κουράγιο. Θα δώσω τώρα εν συντομία το λόγο στους προσκεκλημένους μας από την Ινδονησία. Έχουμε το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθεκτικότητος από την Δημοκρατία της Ινδονησίας και ο διοικητής αυτού του Ινστιτούτου, νομίζω ότι αυτός είναι ο τίτλος σας, θέλετε να μας παρουσιάσετε τον φορέα σας. Παρακαλώ κύριε Κυβερνήτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευκαιρία για μένα να μιλήσω γαλλικά, μια και εσείς είστε Γάλλος. Κρίμα που δεν μπορώ να μιλήσω Ινδονησιακά, δεν έχετε όμως μετάφραση, δεν έχετε διευμηνία. Σας ευχαριστώ καταρχήν Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το κτίριο, το κοινοβούλιο σας. Γιατί ο εκδημοκρατισμός στη χώρα μας ξεκίνησε από το 1998 μετά την πτώση του Σουχάρτο. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε ως ακροατές. Ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ τον πρέσβη και ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές. Έχουμε λοιπόν την Εθνική Αντιπροσωπεία από το Ινστιτούτο αυτό Αντοχής. Οι εκπρόσωποι, τα μέλη εδώ είναι πολιτικοί, αλλά υπάρχουν και ε, αστυνομικοί και στρατιωτικοί Είμαστε σε φάση αποκέντρωσης της ε, εξουσίας της ε, Τζακάρτας. Και επομένως είμαστε σε φάση έτσι εκδημοκρατισμού και αποκέντρωσης της Ινδονησίας. Έχουμε λοιπόν εδώ την οργάνωση αυτή, η οποία είναι μια μη κυβερνητική, επίσης και μια μη κυβερνητική οργάνωση, Υπάρχει λοιπόν και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ο στόχος της αποστολής μας εδώ στις Βρυξέλλες είναι να γνωρίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς μάθατε για μας Στην Ινδονησία, μετά την βόμβα που έσκασε στον Παλί το 2002, άλλαξαν τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα στην ε, Ινδονησία. Υπήρξε ένας, ε, μια ριζοσπαστικοποίηση. Θα ήθελα να μάθω πώς ε, λειτουργεί το δίκαιο εδώ. Τι μέτρα έχετε προβλέψει για το, τις ακραίες ομάδες. Γιατί τα ρωτάω αυτά τώρα. Η παρουσία μας εδώ είναι να κάνουμε μια στρατηγική μελέτη. Ε, έχουμε εδώ ανώτατους υπαλλήλους στους κόλπους μας και θέλουν να μελετήσουν αυτές τις ε, διαφορές. Ο στόχος του Ινστιτούτου μας είναι να παίξει το ρόλο του think tank, του συμβούλου, ας πούμε, του γραφείου του, Προέδρου. Θέλουμε να μάθουμε, λοιπόν, ε, τι στάση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις ριζοσπαστικο... Ε, ομάδες. Ε, εσείς... Και εσείς όπως και εμείς ε, είμαστε μεγάλη χώρα, ε, έχουμε πολλές γλώσσες, έχουμε περίπου 140 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτά θέλω να μάθω και σε ευχαριστώ για την ε, υποδοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας συγχαίρω για τα γαλλικά σας. Δεν είναι εύκολα. Σας ευχαριστώ που μας επισκεφθήκατε. Για το θέμα που, απασχολεί, που σας απασχολεί. Μιλήσατε για την απορριζοσπαστικοποίηση. Δηλαδή εννοείται την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εκτρεμισμού. Κοιτάξτε, οι τρομοκράτες ε, επιτίθενται με όπλα. Υπάρχουν όμως και ορισμένε ομάδες που δεν είναι τρομοκράτες στον πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά έχουν ριζοσπαστικές έτσι, τάσεις και ιδεολογία. Είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε. Ίσως έχετε σχετική εμπειρία. Τι προβλέπει ο νόμος και πώς οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι βουλευτές προωθούν την απορριζοσπαστικοποίηση σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο εκπαίδευσης, ε, ε, οτιδήποτε μέτρο έχετε προβλέψει, οτιδήποτε υπάρχει στην Ευρώπη θα ήθελα να το μάθω. Ο τεράστιο το θέμα και δυστυχώς την απάντηση δεν μπορούμε να σας τη δώσουμε εδώ στην υποεπιτροπή μας. Καταρχάς, ε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση, τα θεσμικά όργανα που θα επισκεφτείτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είσαστε σήμερα εδώ, ε, βασίστηκαν σε αυτή τη διαδικασία από ριζοσπαστικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε από ένα σχέδιο ειρήνης, προσπάθεια ειρήνης της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Το στίχημα, ας πούμε, είναι η ειρήνη μεταξύ των κρατών που επί αιώνες ε, πολέμησαν σε αυτήν εδώ την Υπηρό μας. Είναι λοιπόν μια, ένα εγχείρημα που βασίζεται στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού ε, εναντίον των κινημάτων αυτών των ριζοσπαστικών και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ουσιαστικά ε, είναι σημεοφόροι αυτών των αξιών. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, τι προβλέπει η νομοθεσία. Κάθε κράτος μέλος είναι κυρίαρχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε θέματα νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας Κάθε κράτος έχει τις ιδιαιτερότητές του, ε, έχει το δικό του πλωστάσιο νομοθετικής φύσεως, ούτως υπήν, για να καταπολεμήσει ε, τα εξτρεμιστικά διολυστήματα. Έχουμε τώρα και μια Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ σημαντική επιτροπή, η οποία ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο το γενικότερο και τις συστάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σεβασμό των δικαιωμάτων, των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών, με βάση κάποιες αρχές ε, καθολικές ε, που αναγνωρίζονται και δέχονται όλοι. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να τις προωθήσουμε αυτές τις αρχές ε, παγκόσμια. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις βεβαίως ευρωπαϊκές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ποινικό δίκαιο και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ε, θεσμικό όργανο, ένα δικαστήριο που αποτελεί αν θέλετε, ένα είδος εφετείου σε σχέση με τα εθνικά δικαστήρια και σε σχέση με τις δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάποια εθνικά δίκαια. Μπορεί να προσφύγει κανείς λοιπόν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά τελεσίδικα και αυτό είναι τμήμα, ας πούμε, της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Ε, θέλω να έρθετε σε επαφή με τα μέλη, με τους βουλευτές, δηλαδή, της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, όπως τη λέμε, για να δείτε ε, μέσα σε ποιο πλαίσιο δουλεύουν, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν αυτή τη μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ε, νομοθεσιών, των εθνικών νομοθεσιών, δηλαδή. Επίσης, για, σε πιο τεχνικό επίπεδο έχουμε και ένα συντονιστή για την καταπολέμηση τρομοκρατίας ε, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, εξωτερική δράση, ένα νέο θεσμικό όργανο και αυτό ο συντονιστή έχει ένα πιο ταπεινό ρόλο. Δεν υπάρχει μία ευρωπαϊκή πολιτική κατά της τρομοκρατίας. Υπάρχει μια στρατηγική ευρωπαϊκή, ναι, κατά πολέμηση της τρομοκρατία. υπαρχει μια στρατηγικη ευρωπαικη ναι κατα πολεμηση τη τρομοκρατία και μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, όπου εκεί εντάσσεται η καταπολέμηση τη τρομοκρατία ω προτεραιότητα, αλλά παρόλα αυτά τα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα έχουν ε, τα δικά τους όπλα, έχουν τις δικές τους διατάξεις, έχουν διαφορετικό δυναμικό καθένα, ανάλογα με το μέγεθος, ανάλογα με τη γεωγραφία τους, ανάλογα με την εμπειρία και την ιστορία τους ε, και τη σχέση με αυτά τα τρομοκρατικά και ριζοσπαστικά φαινόμενα. Εδώ τώρα στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας ασχολούμαστε, όπως ακούσατε προηγουμένως, ε, με την παρακολούθηση κάποιων εξωτερικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη στρατιωτικέ όπω ακούσατε. Σήμερα το πρωί έχουμε 8 τέτοιε αποστολέ, αλλά και στρατιωτικέ αποστολέ. Έχουμε τρει στρατιωτικέ αποστολέ αυτή τη στιγμή, εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό τη επικράτησης Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ο ρόλο τη υποεπιτροπή στην οποία βρισκόσαστε. Αυτό δεν μα απαγορεύει βεβαίω να έρθουμε σε επαφή με του υπεύθυνου ε, για θέματα τρομοκρατία, ε, να, μιλήσουν όμως ε, για θέματα ασφάλειας περισσότερο, όχι για θέματα νομοθεσίας για την τρομοκρατία, έτσι, για τέτοια θέματα μας μιλάνε. Θέματα ασφάλειας. Ε, αυτά έχω να σας πω εγώ. Ίσως κάποιος μπορεί να με συμπληρώσει. Ο κύριος Γκάλερ, η κυρία Νέιτς. Να καλωσορίσω την τόσο σημαντική Ινδονησιακή αυτή αντιπροσωπεία, θα ήθελα, διότι ο σύζυγός μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε αρκετά και να επισκεφτούμε την Ινδονησία. Όχι βεβαίω όλη την Ινδονησία, γιατί η χώρα σας είναι τόσο μεγάλη, τεράστια. Και θα ήθελα να χαιρετήσω την προσπάθεια που καταβάλουν οι Ινδονησιακές αρχές, εδώ και πολλά έτη μάλιστα, προκειμένου να καταπολεμήσουν αυτή την ριζοσπαστικοποίηση. Διότι κατάλαβαν τι κίνδυνο συνιστά και απειλεί καταρχήν τους ίδιους τους Ινδονήσιους. Ελπίζω συνεπώς ότι κατά διάρκεια της ε, εδώ παραμονής σας στις Βρυξέλλες θα έχετε μια ανταλλαγή εμπειριών η οποία νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για σας. Αν θα μπορούσα και εγώ να πω κάτι, να προσθέσω ότι η Ινδονησία είναι μία από τις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπειρία, αν θέλετε, εξωτερικών επιχειρήσεων. Διότι είχαμε και μια επιχείρηση, αν θέλετε, διαμεσολάβησης, η οποία απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμη. Για πρώτη φορά έγινε μια τέτοια αποστολή τόσο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδε η Ινδονησία δηλαδή πόσο προσιλωμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαδικασίες, αν θέλετε, διαμεσολάβησης. Κύριε Κυβερνήτα, αν έχετε κάτι να προσθέσετε, σας ευχαριστώ. Για λογαριασμό εκ μέρου ε, και της ε, Ινδονησιακής κυβερνήσεως. Και κατάλαβα τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη σχέση αυτής της αποστολής. Όπω επίση και στην αντιμετώπιση, αν θέλετε, του προβλήματος που δημιουργήθηκε με το τσουνάμι. Γιατί αυτό σημαίνει ανθρωπισμός. Πολλοί Ινδονήσιοι πιστεύουν ότι οι Ευρωπαίοι βοηθούν πάρα πολύ. Ξέχασα βεβαίως να σας πω προηγουμένως να πω ότι ευχαριστώ όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ κύριε Κυβερνήτα για τα ευγενικά σας λόγια Είστε ευπρόσδεκτοι για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα εύχομαι αν θέλετε μια γόνιμη, πραγματικά καρπερή αν θέλετε και καλή διαμονή σας εύχομαι. Εδώ ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας. Θα ξαναβρεθούμε στις 12 Ιουλίου για την ακρόση της αποστολής, αν θέλετε, στην Δημοκρατία του Κονγκό.